Μια και δεν υπάρχουν, ε, αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις ε, για τα πρακτικά, θα, μεταβλη, ε, θα, διαβιβαστούν τα έγγραφα σε όλα τα θεσμικά όργανα που αναφέρονται, αναφέρονται στο, στην ημερήσια διάταξη. Διακοπή της Συνόδου, καλό απόγευμα και καλό ταξίδι.